Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινήσουμε σε ένα λεπτό τη συνεδρίαση και σας παρακαλώ να καθίσετε. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu. Άρχεται η συνεδρία σας κηρύσω την ε, επανέναρξη της ε, περίοδου συνόδου που είχε διακοπεί στις 11 Νοεμβρίου. Τα κείμενα που έχουν υιοθετηθεί καθώς ε, και τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 11 Νοεμβρίου είναι στη σας. Δεν βλέπω παρατηρήσεις. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά. Ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις καταρχάς. Με μεγάλη ικανοποίηση ενημερωθήκαμε ότι η κυρία Αουν Σανσουτσί έχει απελευθερωθεί. Πρόκειται βεβαίω για την πολύ γνωστή ηγέτητα τη αντιπολίτευση τη Πυρμανία. Πρόκειται για μία από τι πρώτε πολιτικού, από του πρώτου πολιτικού που τιμήθηκαν με το βραβείο Ζαχάροφ, που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις αγωνιστές της ε, ελευθερίας Συνεδρίου από το 1989. Δυστυχώς δεν έχουμε μπορέσει να την δούμε την ίδια για να τι απονείμουμε, να τις επιδώσουμε το βραβείο αυτό. Εγώ της επέστειλα επιστολή ζητώντας της, εάν έχει την ευκαιρία, να έρθει μέχρι εδώ για να της απονείμουμε το βραβείο σε μια ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 25 Οκτωβρίου έλαβε χώρα, εορτάστηκε μάλλον, η 11η ε, η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Οι γυναίκες καθημερινά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, βιασμών, υποφέρουν με διάφορους τρόπους και από διάφορους μορφές καταπίεσης οι γυναίκες. Είναι πολύ υψηλά τα νούμερα των νέων κοριτσιών που θύματα βιασμού κάθε χρόνο και θέλοντας να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτές τις βαρβαρότητες, καταθέτουμε και καταγράφουμε τις, ε, ε, τη βούλησή μας για να περατωθεί κάθε μορφή φυσικής ή ψυχολογικής βίας της βάρος των γυναικών. Άλλε ανακοινώσει. Οι αρμόδιε Ισπανικέ Αρχέ με ενημέρωσαν ότι ο κύριο Ραμόν Χαουρεγκούι Ατόντο αντικαθίσταται από την κυρία Μαρία Ιριγκοϊέν Πέρες από 16 Νοεμβρίου του 2010. Καλώς ορίζω τη νέα συνάδελφο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι. Υπενθυμίζω δε ότι δυνάμει το άρθρο 3 παραγραφός 2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο δεν έχουν επαληθευθεί ε, οι συνθήκες εκλογής ή όσο δεν έχει γίνει επαλήθευση ενδεχόμενης ένστασης, η κυρία Μαρία Ιριγκόιεν Πέρες, ε, εδρεύει μέσα στο κοινοβούλιο και στα λοιπά του όργανα, έχοντας πλήρη δυνατότητα άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι έχει εντωμεταξύ καταθέσει τη δήλωση πως δεν ασκεί δραστηριότητα ασύμβατη με το λειτουργήμα του Ευρωβουλευτή. Επίση, θέλω να σα ενημερώσω ότι ο κύριος Κλάουδιος Σύπριαν προσχώρησε στην ομάδα της προοδευτική Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 15 Νοεμβρίου του 2010. Σα ενημερώνω επίσης πως ο κύριος Πίνο Αρλάκη προσχώρησε στην ομάδα της προοδευτική Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 18 Νοεμβρίου του 2010. υπογραφή πράξεων που υιοθετούνται υπό τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με τον πρόεδρο του Συμβουλίου πρόκειται να ε, συνυπογράψουμε 14 ε, πράξεις νομοθετικές που υιοθετήθηκαν υπό τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ε, δυνάμει του άρθρου 74 του κανονισμού του Κοινοβουλίου και θα δημοσιευθούν οι πράξεις αυτές στα πρακτικά της περίοδου συνόδου ε, της παρούς περίοδου συνόδου είναι στη διάθεσή σας για ενημέρωση και πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή. Τώρα προχωρώ στις τροποποιήσεις της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου, δυνάμει το άρθρο 137 του κανονισμού. Για τη Δευτέρα, γιατί θα κοιτάξουμε κάθε μέρα με τη σειρά από την ημερήσια διάταξη. Στη Δευτέρα λοιπόν οι πολιτικές ομάδες προτείνουν η συζήτηση για την έκθεση του κ. Μπερλενγκουέρ ως προς τις ε, πτυχές του προγράμματος δράσεως εφαρμογής του προγράμματος Στοκχόλμης επί του αστικού εμπορικού οικογενειακού και διεθνούς και δικαίου ε, να φύγει από την ημερήσια διάταξη, να μην ε, συζητηθεί στην ημερήσια διάταξη και θα, να ψηφιστεί απευθείας αύριο. Θα εξεταστεί λοιπόν η έκθεση αυτή, αλλά χωρίς συζήτηση, μόνο με ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω. Μας ενημέρωσαν όλες τις πολιτικές ε, ομάδες ότι την πρόταση αυτή, η έκθεση Berlinguer, να μην ε, συζητηθεί και να περάσει απευθεία ψηφοφορία, τις ε, βρίσκει όλες σύμφωνες. Για την τρίτη δεν έχουμε καμία τροποποίηση. Κύριε Σούλτς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, για την τρίτη η μερίσια διάταξη αναφέρεται σε έξι εκθέσεις του κυρίου Ματέρα, της κυρίας διορθώνει ο για τη χρήση του ε, Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, για την ε, αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης υπέρ των κατοχωρών. Θα ήθελα να λάβω το λόγο γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο σφάλμα το ότι ο κύριος Ντόλι πέστη τα πυρά του ε, Ολλανδικού τύπου ε, για ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στη διάσκεψη των Προέδρων, όπου ετέθη ζήτημα εάν η έκθεση αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει τη συζήτηση για τον προπολογισμό ή μη. Θα ήθελα λοιπόν να κατήσω σαφέ ότι θα πρέπει να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη έκθεση μάτερα ότι θα πρέπει να συζητηθεί, να ψηφιστεί και να μεταφερθούν τα σχετικά κονδύλια από το Τομείο Παγκοσμιοποίηση, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Πρώτον. Δεύτερον όμω, έγινε μία παρατήρηση στη των Προέδρων, η οποία θα έπρεπε ή μη τι άλλο να του επιτρέψει να κάνει δηλώσεις ή επεξηγήσεις για τα όσα ε, υπόθηκαν. Δηλαδή να μην ε, πιέζεται κανείς εάν δεν έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει την τοποθέτησή του. Εδώ δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι κάτω χώρες ή μάλλον το κοινοβούλιο δα, ε, ξοδεύει λεφτά, πετάει λεφτά από το παράθυρο. Οι κατοχώρες είναι αυτές που κατηγορούν το Κοινοβούλιο πως έχει μια τέτοια ανεύθυνη πράξη. Όμως η κυρία Ματέρα έχει μια πολύ υπεύθυνη στάση στην υπόθεση αυτή και πιστεύω ότι η έγκριση της διάθεσης των σχετικών κονδυλίων ε, από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης αποδεικνύει ακριβώς ότι είμαστε υπεύθυνοι και με πολύ μεγάλη σύνεση διαθέτουμε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ. Ξέρω. Ξέρω το ζήτημα αυτό. Γνωρίζω επίσης ε, και τα διάφορα άρθρα που αναφέρθηκαν στον Ολλανδικό τύπο. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι τα σημεία αυτά για την κινητοποίηση του, Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση παραμένει στη μερίσια διάταξη και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Δεν αλλάζει τίποτα. Κυρίε και κύριοι, πάμε στην ε, Τετάρτη. Η ε, Ενωτική Αριστερά πρότεινε η συζήτηση για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα να ακολουθηθεί από ψηφοφορία επί προτάσεως ψηφίσματος σχετικά με το θέμα σε αυτή τη σύνοδο και όχι το Δεκέμβριο όπως είχε προγραμματιστεί. Θα ακούσουμε την πρόταση του κυρίου Φερέρα. Κύριος Φερέρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα είναι αρκετά σοβαρή και έτσι το Κοινοβούλιο μας θα πρέπει να τοποθετηθεί γρήγορα επί του θέματος. Ξέρουμε τα γεγονότα ποια είναι. Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει. Είδαμε την καταστροφή των διαφόρων ε, καταβλισμών των κατοίκων της συστικής Σαχάρας, των Σαχαράουι. Εξαφανίστηκαν άνθρωποι, σκοτώθηκαν άνθρωποι, εμποδίστηκαν και ευρωβουλευτές να πάνε εκεί, τους ε, απόθυσαν οι μαροκινές αρχές. Το ίδιο έχει γίνει και με βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων και με δημοσιογράφους και με μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Το να μην τοποθετηθούμε επ' αυτού τώρα ε, θα ήταν ε, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητό και θα ήταν μια στάση απαράδεκτη. Σχεδόν συνενοχή θα αποτελούσε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν αντιπροσωπεύει τι αξίε που προσπαθούμε να προωθήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να λάβετε μια λογική ε, απόφαση και να υποστηρίξετε την ψήφο, την ψήφο αυτού του ψηφίσματος και να υποστηρίξετε την πρότασή μας. Αυτό θα ήθελα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να καλέσω κάποιον που θα ήθελε να μιλήσει υπέρ της προτάσεως αυτής. Υπέρ της προτάσεως αυτής. Τα επιχειρήματα που προευλήθησαν από την ΚΟΕ ε, ε, είναι σωστά, οπότε θα υποστηρίξω αυτή τη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος να μιλήσει κατά της προτάσεις, ο κ. Σούλτς. Πρόεδρε, θα παρακαλώ τον κύριο Φερέρα να μου δώσει την προσοχή του για ένα λεπτό. Στη διάσκεψη των Προέδρων και κατά την προετοιμασία τη διάσκεψη των Προέδρων συζητήσαμε εντατικά το θέμα αυτό και θα ήθελα εκ μέρου τη ομάδα μου να πω ότι ανησυχεί ιδιαίτερα η ομάδα μου για τα εκτενόμενα στη Δυτική Σαχάρα και αν αληθεύουν εικόνα που είδαμε θα πρέπει όχι μόνο να γίνει σοβαρή συζήτηση αλλά ενδεχομένως και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Σοβαρότητα σημαίνει να συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα τα γεγονότα ο Υπουργό των Εξωτερικών όμω του Μαρόκου μα έχει δηλώσει ότι πρόκειται να έρθει στην Επιτροπή των Εξωτερικών. Δεν είναι υποχρεωμένο να το πράξει αυτό. Δεν είναι υποχρεωμένο να έρθει να μιλήσει στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όμω είναι διεθυμένο να το πράξει. Α το αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτό σαν ευκαιρία. Α δούμε εάν ευσταθούν όλε τι κατηγορίε και μετά να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα. Είναι πολύ πιο σοβαρό αυτό από το να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα, να το ψηφίσουμε και μετά να ακούσουμε τον Υπουργό των Εξωτερικών του Μαρόκου. Ας δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Υπάρχει δυνατότητα από πλευρά τη Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων να ακροαστεί τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου και να δει τι έχει να απαντήσει. Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ πιο συνεπή και σοβαρή στάση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε τώρα. Ποιο είναι υπέρ του... τη προτάσεω αυτή. Ποιο είναι υπέρ της προτάσεως του κυρίου Φερέιρα. Σας ευχαριστώ. Ποιος είναι κατά της προτάσεως του κυρίου Φερέιρα. Πρέπει να διεξαχθεί έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος θα λάβει χώρα τώρα. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, εγκρίνεται αυτή η πρόταση. Η πλειοψηφία είναι υπέρ. Έτσι, σύμφωνα με την πρόταση του κυρίου Φερέιρα, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αυτή την εβδομάδα. Και θα σας γνωστοποιήσω το πότε. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Πέμπτη προθεσμίες είναι εξή και προσέξτε σας παρακαλώ. Προτάσεις ψηφίσματος μέχρι το μεσημέρι αύριο, την 3η 23 Νοεμβρίου. Λοιπόν, μεσημέρι αύριο για τις προτάσεις ψηφίσματος. Λοιπόν, προθεσμία για τροπολογίες και κοινέ προτάσεις ψηφίσματος είναι μεσημέρι Τετάρτη, μεθαύριο. Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Αυτή είναι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών και κοινών προτάσεων ψηφίσματος. Και τέλος, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για τι τις προτάσεις ψηφισμάτων είναι στις 1 η ώρα την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, δηλαδή μία ώρα αργότερα. Θα το επαναλάβω. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ δεν προτάθηκαν κάποιες αλλαγές για την Πέμπτη και η ημερήσια διάταξη αυτής της Συνόδου θεωρείται ως εγκεκριμένη. Θα ήθελα να, ζητήσω από, να ρωτήσω τους συναδέλφους κάτι. Υπάρχει ένα κατεπήγον όσον αφορά τη, το Θιβέτ την Πέμπτη και ότι η Κίνα θέλει να επιβάλλει την κινέζικη γλώσσα στο Θιβέτ. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρήζει συζητήσεως στην Ολομέλεια, παρουσία της κυρίας Άστον. Δεν είναι απλώς ένα θέμα κατεπήγων. Μιλάμε για τη θεμελιώδη πολιτική της Κίνας αυτή τη στιγμή που την ασκεί στο Θιβέτ και νομίζω ότι ξεπερνάει το θέμα των κατεπηγόντων. Ε, ε, εντάξει, το κατεπήγων καλώς αν το επιθυμεί η πλειοψηφία. Και εγώ αν είναι δυνατόν και ξέρω ότι η μερίσια διάταξη δεν είναι τόσο γεμάτη το Δεκέμβριο αν μπορούμε να το εξετάσουμε το θέμα μετασυζητήσεως και μεταψηφίσματος και παρουσία της κυρίας Άστον όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έναντι της Κίνας, όσον αφορά αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ ενδειγμένο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, κύριε Κονβέντιτ. Να το θέσετε αυτό, σας παρακαλώ, στη διάσκεψη των Προέδρων, ελεύθερα. Σαν Πρόεδρος της πολιτικής σας ομάδας έχετε αυτή τη δυνατότητα. Σας ευχαριστώ.